No, no, no, no, no, no, no. La seduta è aperta. Συνεχίζεται τη συνεδρίαση. Πριν απευθύνω χαιρετισμό στον Επίτροπο, ο κύριος Βέμπερ έχει στήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για ένα κατεπήγον θέμα. Αυτό το οποίο γύρετε και εσείς με τη δική σας δηλώση χθες, τη δολοφονία της βάρος του Σλοβάκου δημοσιογράφου. Σήμερα ακούστηκαν νέες πληροφορίες από τη μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα ακόμα δύο δημοσιογράφοι φαίνεται να έχουν δολοφονηθεί μετά τη δολοφονία στην ε, Μάλτα και το, η Σλοβακία. Ε, θα σας παρακαλέσω λοιπόν, ε, μια και δεν υπάρχει ακόμη διάσκεψη στον Πρόεδρο αυτή την εβδομάδα, δεν προβλέπεται άλλη συνεδρίαση, να ε, αναλυφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαρευνηθεί πλήρως αυτό το έγκλημα, αυτά τα έγκληματα και βεβαίως να ε, ληφθεί και μέρημνα ώστε να εξεταστεί αν τυχόν κονδύλια ευρωπαϊκά έχουν τύχει κατά ε, χρήσεως να αποσταλεί μια ε, ομάδα βουλευτών ως αποστολή διερευνητική στη Σλοβακία. Πρέπει το, φως να το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ο φανός εκείνος ο οποίος θα φωτίσει το σκοτάδι της διαφθοράς και θα αποκαλύψει τα εγκλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούλμαν. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το κοινοβούλιο μας, και το λέω εξ της ομάδας μου, δεν έχει να πάρει μαθήματα από κανέναν στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και στη διερεύνηση και διελεύκανση ε, ανεπιφύλακτα όλων των εγκλημάτων και των παραβιάσεων. Γι' αυτό, εάν το επιτρέπει η κατάσταση, να κάνουμε συζήτηση. Είμαστε υπέρ, νομίζω είναι συνένεση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω ότι η αποστολή που προτάθηκε από τον συνάδελφο Βέμπερ είναι στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής τάξη Δηλαδή προβλέπεται για τη νέα Εξεταστική Επιτροπή που θέλουμε σήμερα να στήσουμε και θα παρακαλέσω να έρθετε σε επαφή, ε, Πρόεδρε, με τους ε, αρμοδίους στην Επιτροπή Τάξη 3 για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Κατά τα άλλα θέλω να θυμίσω στον κύριο Βέβε ότι θέλουμε να χεθεί άπλετο φως, χωρίς καμία επιφύλαξη, ανεξαρτήτως κράτους μέλους, ανεξαρτήτως ε, της εκάστοτε κυβέρνησης, μπορεί να είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κάπου, πούμε, δεν θα μας εμποδίσει αυτό να το διαρευνήσουμε με τρόπο ξεκάθαρο ε, και αυτό αφορά και πρόσφατα σκάνδαλα διαφθοράς, καταγγελίες, σε βάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Bene. Ruiz. Thank uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω ότι φόνοι δημοσιογράφων δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικών πολιτικών. Είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα. Το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πολύ σκληρή δράση με την δολοφονία στη Μάλτα. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ένα τέτοιο έγκλημα συμβαίνει στη Σλοβακία. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση του κυρίου Βέμπερ για αποστολή μιας ειδική ομάδας στην Σλοβακία και επί τη ευκαιρία Παρακαλώ αυτό να γίνει με εντολή τη έσκεψη των Προέδρων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να περάσουν μερικέ εβδομάδε μέχρι ότου συσταθεί η νέα γραμματεία για τη νέα επιτροπή. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δρουν ελεύθερα ακόμα και όταν διερευνούν θέματα διαφθορά και φοροδιαφυγή. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Σα ευχαριστώ. Sono ο Πρόεδρος, είμαι και εγώ πεπισμένος ότι η ελευθερία του τύπου δεν είναι θέμα ούτε της αριστεράς, ούτε της δεξιάς, ούτε του κέντρου. Η ελευθερία του τύπου είναι αξία θεμελιώδης για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να είναι θεμελιώδης για κάθε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πολιτικής χρειάς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι να ε, ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία γραπτή συνεννόηση μεταξύ των Προέδρων των πολιτικών ομάδων προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για αποστολή μια ομάδα βουλευτών και αναλόγω θα, θα, θα διαθετήσουμε το τυπικό θέμα στην Σλοβακία για να μελετήσει, να ερευνήσει τι έχει συμβεί, όπω άλλωστε έχει συμβεί και με τη Μάλτα. Προτείνω λοιπόν γραπτή διαδικασία να ξεκινήσει το απόγευμα, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σήμερα συνελήφθησαν δυστυχώς επιτρέψτε μου συνελήφθησαν δυστυχώς τρεις Ιταλοί πολίτες που ζούσαν στην Σλοβακία. Ωστόσο πρέπει να αντιληφθούμε όχι μόνο ποιοι είναι οι αυτούργοι αλλά πάνω απ' όλα οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας. Όπως άλλωστε πρέπει να αναζητηθούν οι ηθικοί αυτούργοι της Ντάφνη Καρουάνα. Εγώ σε αυτό θα συνεχίσω να επιμένω. Δεν μπορούμε να δίνουμε μαθήματα σε άλλους εάν δεν ε, καθαρίσουμε τα του οίκου μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή η διαδικασία. Όπως είπα, γραπτός ξεκινάει η διαδικασία. Θα μπορέσουν όλες οι πολιτικές ομάδες να εκδηλώσουν βούληση και προτιμήσεις για να αποσταλεί το ταχύτερο δυνατό αυτή η ομάδα. Η κυρία Μουσολίνη έχει το λόγο, πρόεδρε ομιλώ και εκ μέρους του Αλμπέρτο Σιτσίριο για την ε, Σλοβακία. Λοιπόν, εμείς πρόκειται να καταθέσουμε μια προφορική ερώτηση. Είπε ο κύριος Βέμπερ ότι μπορεί να υπάρχει κατάχρηση κονδυλίων, μα υπάρχει κατάχρηση ακόμα και του εσωτερικού ντάμπινγκ και αναφέρομαι εδώ στους ε, εργαζομένους που πρόκειται να απολυθούν από μια εταιρεία η οποία από την Ιταλία μετακομίζει στη Σλοβακία. Πρόκειται για μια ε, πρακτική απαράδεκτη που δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος είναι ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Προσωπικώ ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Ε, χθες ακόμη, συνοδευόμενος και από τον ε, πρόεδρο της, ε, του Πεδεμοντίου, είχα συνάντηση με τους συνδικαλιστές εκπροσώπους ε, των εργαζομένων αυτής της επιχείρησης ε, και έχω δεσμευθεί για μια συγκεκριμένη απάντηση. Είμαι λοιπόν σε επαφή με τα συνδικάτα, τον πρόεδρο της, ε, τον Περιφερειάρχη, αλλά και την κυβέρνηση της Θελής, κυρία για πρώτα, αλλά όχι. Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μιλάτε για τα κράτη-μέλη και την τήρηση του κράτους δικαίου. Μιλάτε για δολοφονίες εις βάρος δημοσιογράφων. Ο κύριος Μούσνιακ είναι εδώ και θα απευθυνθεί στο σώμα. Νομίζω ότι είναι η ώρα να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε τον Πατ Φανούκα, αγωνιστή δικηγόρο, αγωνιστή των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ο οποίος ξέρουμε το δολοφονήθηκε από εκπροσώπους των Unionists με κάποια συμπαιχνία και της κυβέρνησης της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Ε, ήρθε η ώρα λοιπόν να μνημονεύσουμε και αυτή τη δολοφονία. Κυρία Τόγια έχει το λόγο. Γνωρίζουμε, εκτιμούμε ιδιαίτερω αυτά τα οποία πράξατε χθε, Πρόεδρε, την πρωτοβουλία σα και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν ε, αποτελέσματα ουσιαστικά σε παιδοκυβέρνηση κυβέρνηση τη Ιταλία. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουμε από τι πολυεθνικέ που έχουν και κοινωνική ευθύνη ε, όταν καταθίστανται σε μια χώρα, αναπτύσσουν δραστηριότητες, δίνουν θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να τα κλείνουν, να κλείνουν τις εγκαταστάσεις ε, για, το λόγο αυτό, για απλούς λόγους οικονομικής αξιολόγησης. Πρέπει λοιπόν να γίνει μελέτη και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά και με κάθε άλλο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι ευρωπαϊκά ε, κονδύλια, περιφερειακά κονδύλια και ταμεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη κάποιων περιφερειών να μην χρησιμοποιούνται για λόγους κοινωνικού ντάμπινγκ, για λόγους έργασία του ντάμπινγκ. Θα πρέπει να διερευνηθεί αυτή η επιχείρηση λοιπόν για κάθε κονδύλιο που έχει λάβει από ευρωπαϊκούς πόρους και για τον τρόπο με τον οποίο τα έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος. Καλώς και ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, Έχω την τιμή να ηγούμε ε, τη αποστολή στη Μάλτα και ε, θέλω να συμφωνήσω πως όντως πολλή δουλειά πρέπει ακόμα να γίνει. Ε, περιμένουμε απάντηση από εκεί, όμως η δουλειά που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να γίνει μέσα στην εντολή της νέας επιτροπής που θα φτιαχτεί. Ε, μιλήσαμε όμως και για την κυρία Μογκερίνη. Θέλουμε να ρωτήσουμε μάλλον την κυρία Μογκερίνη για την κατάσταση στην Αιθιοπία. Έχει παρατηθεί ο πρόεδρος, υπάρχει η κατάσταση επίγουσας ανάγκης και η κατάσταση, η θέση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι ντροπιαστική. Ε, οι Αμερικανοί ήδη κατέ, καταδίκασαν ε, τις εξελίξεις εκεί και σε ζητώ να φτιάξουμε μια θέση που να σέβεται τις αξίες μας και να ανταποκρίνεται στα ε, δημοκρατικά μας ε, πρότυπα για το τι συμβαίνει στην Αιθιοπία και την κατάσταση του κράτου δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνουμε συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητήσατε τον λόγο για επίγοντα θέματα, αλλά έχουμε και έναν φιλοξενούμενο και είναι καθήκον μας. Μπορούμε να παρέμβουμε πριν από τη συζήτηση γιατί πράγμα θέλετε το λόγο κυρία Άρμασα Εγώ θέλω να σας ζητήσω Πρόεδρε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη διότι για το θέμα που συζητάμε ε, καλό είναι να ακούσουμε τον ε, κύριο Νιεσταμουνούτσνικτ. Ε, ναι, αυτό θα κάνουμε. Αλλά υπόθεση του δολοφονημένου ε, δημοσιογράφου είναι τόσο σοβαρή υπόθεση που και η Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που του καλέσαμε, την καλέσαμε η κυρία Βυσνιέσκα κατάλαβε πολύ καλά ποια είναι η σημασία του θέματος και την ευχαριστώ, ε, την ευχαριστώ που ε, έκανε υπομονή για λίγα λεπτά γιατί και αυτό ήταν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας καλωσορίζω. Εσείς είστε επίτροπος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς συμμεριζόμαστε την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων και ε, θέλουμε να μιλήσουμε για την ε, βία κατά των γυναικών και την και, οικογενειακή